εξωτερική πολιτική, την κυρία Μογκερίνη, θα μας μιλήσει για την κατάσταση στη Συρία. Έχετε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι συζητήσαμε το θέμα στη Συρία. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τερματιστεί ο πόλεμος στις 19 Ιανουαρίου, λιγότερο από δύο μήνες από τότε έχουν μεσολαβήσει πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω λοιπόν για τη συζήτηση που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε σήμερα για να ελέγξουμε τα βήματα τα οποία έχουν γίνει, να ελέγξουμε την κατεύθυνση την οποία έχουμε ακολουθήσει και τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει συμβεί μέσα σε αυτόν τον 1,5 μήνα Καταρχάς έγινε η διάσκεψη του Λονδίνου, ξεκινώ από αυτό, γιατί αυτό δεν ήταν μόνο δωρητές και δωρήτριες που εκπροσωπήθηκαν εκεί. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί τα δύο τρίτα των πιστώσεων για τη στήριξη των σύρων στο εσωτερικό και στις ε, γύρω χώρες αλλά ταυτόχρονα απέδειξε την ενότητα τη διεθνούς κοινότητας και ε, θα έλεγα ταυτόχρονα έδειξε ε, και μια κάποια ελπίδα για τους Σύρους, τρία δις ε, κατευθύνονται προς την κατεύθυνση αυτή και στο εσωτερικό της Συρίας και στις όμορες χώρες και θα επανέλθω στο θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο ασφαλείας. Προετοιμάσαμε επίσης δύο κόμπαξ, δύο πακέτα, ένα για το Λίβανο και ένα για την Ιορδανία που αποτελούνται όχι μόνο από χρηματοδοτικές ε, ε, βοήθειες αλλά και από επιμέρους μέτρα που θα στηρίξουν τις χώρες αυτές στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των σύρων προσφύγων ε, στις κοινότητες που τους φιλοξενούν στα πλαίσια της εκπαίδευσης, παιδείας, ευκαιριών για την εργασία και καθιστώντας για τις ίδιες τις κοινότητες τις τοπικές στο Λίβανο και στην Ιορδανία να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αυτές μέσω πρόθεσμα. Το δεύτερο που συνέβη από τις 19 Ιανουαρίου είναι ότι έγινε, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στους Σύρους. Διακόπη σχεδόν άμεσα, διότι ήταν σαφές τα ποια ήταν τα προβλήματα τα οποία ήρθαν στην επικαιρότητα υπό την καθοδήγηση του κ. Ντεμιστούρα και ταυτόχρονα υπήρξε συνάντηση της ομάδας στήριξης στην, στο Μόναχο υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών, τον Κέρι, τον Λαυρόφ, υπήρξαν εκπρόσωποι 20 χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά, προσπαθώντας ακριβώς να δουν τους τρόπους με τους οποίους η διακοπή των συνομιλιών στην Γενέβη οφείλεται σε δυσκολίες οι οποίες είναι ανέφικτο να ξεπεραστούν όχι μόνο εθνικά εσωτερικά στη Συρία αλλά και στο ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο ή μήπω θα ήταν δυνατόν μέσω της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης να υπάρξουν κάποια βήματα προς τα εμπρός και να ε, υπάρξει εκ νέου ε, μια ζωτική όθηση στην προσπάθεια που τόσο χρειαζόμαστε όλοι. Μετά από τη συνάντηση του Μονάχου δημιουργήθηκαν δύο task force. Η μία αφορά τους τρόπους ε, κατάπαυσης του πυρός, προεδρεύεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ρωσία που είναι οι δύο εταίροι οι οποίοι απαιτείται να συντονιστούν σε επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας και να βρούνε ακριβώς ε, με συγκεκριμένο τρόπο την γεωγραφική κάλυψη της χώρας στην οποία ε, θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Και από την άλλη δημιουργήθηκε η Task Force για ανθρωπιστική βοήθεια γιατί εντοπίστηκε η ανάγκη να υπάρξουν ε, διαπραγματεύσεις σε ένα επίπεδο δευτέρου επίπεδου που τις ανακοίνωσε ίδιο ο Στεφάντε Μιστούρα για τις επόμενες ημέρες αλλά σε ένα εντελώς διαφορετικό, πολύ διαφορετικό πλαίσιο στη Συρία σε σχέση με αυτό το οποίο βιώσαμε την προηγούμενη φορά. Τι εννοώ με αυτό. Να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις διαφορές ανάμεσα στους Σύρους που συνομιλούν στην Γενέβη, μια πολύ δύσκολη πολιτική διαδικασία και να υπάρχουν θάνατοι συνεχείς από την άλλη στο εσωτερικό της Συρίας. Ξέρουμε λοιπόν ότι ε, προσπαθούμε να δώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα, φάρμακα στους ήρους στο εσωτερικό της χώρας. Αν το πετύχουμε αυτό δημιουργείται μια αξιόπιστη διαδικασία ειρηνευτικών συνομιλιών στην Γενέβη και ταυτόχρονα ανοίγουν και κάποιες ε, πολιτικές συζητήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στη σύραξη. Λαμβάνοντας αυτά όλα υπόψη λοιπόν, Γνωρίζετε ότι η Task Force ε, για την κατάπαυση του πυρών έχει προχωρήσει, έχει ε, πολλά απτά αποτελέσματα, το ίδιο και σε επίπεδο ε, της Task Force για την ανθρωπιστική βοήθεια όπως και το 2266 ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Από τότε θα ήθελα να πω και δεν το λέω μόνον εγώ αυτό αλλά και ο Στεφάντε Μιστούρα όπως επίσης και οι δύο συμπρόεδροι της Task Force, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία, ότι η κατάπαυση του πυρός εν πολλής κρατή έχουν υπάρξει αρκετές παραβιάσεις σε διάφορα σημεία της Συρίας σε διαφορετικά σημεία της Συρίας. Όμως ε, νομίζουμε ότι η συμφωνία γίνεται εν πολύ σεβαστή η κατάσταση αυτή την εβδομάδα που προηγήθηκε έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες της ενόπλης σύραξης. δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, ή η πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια συνεχώς, συνεχούς σύραξης δεν έχουν υπάρξει ε, μεγάλες σε μέγεθος στρατιωτικές συγκρούσεις. Βέβαια παραβιάσεις επιμέρους υπάρχουν, αλλά σε μια διαφορετική κλίμακα από ό,τι στο παρελθόν. Πάντα στα πλαίσια της Task για την ανθρωπιστική βοήθεια πετύχαμε τις τελευταίες εβδομάδες να παραδώσουμε βοήθεια με 180 φορτηγά σε 185 σύρους στο εσωτερικό της χώρας συνεργαζόμενοι με τα Ηνωμένα Έθνη και θα επανέλθω σε αυτό προσπαθώντας να φτάσουμε σε περιοχές οι οποίες είναι πέραν αυτών στις οποίες έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Όπως είπα επίσης ο Στεφάντη Μιστούρα είπε ότι από αύριο θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Δεν νομίζω ότι θα είναι μια εύκολη διαδικασία, αντίθετα. Όμως είναι καλό το ότι ο Ντιμιστούρα κατάφερε να δημιουργήσει εκ νέου ή όχι θα δούμε τις συνθήκες έτσι ώστε να ξεκινήσουν πάντα οι συνομιλίες. Εγώ συναντήθηκα με ορισμένους από τους εμπλεκομένους στο Παρίσι πριν από ορισμένες μέρες ε, μου είπε ότι δεν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για την επιστροφή ε, στις συνομιλίες αλλά παρόλα αυτά η διεθνής κοινότητα έχει βοηθήσει τις ίδιες τις συνομιλίες ε, να αποκτήσουν περιεχόμενο. Και ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να αποστείλουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα είναι να ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές το ίδιο το καθεστώς και την αντιπολίτευση επίσης να πάνε στη Γενέβη και να, να μπορέσουν να εμπλακούν σε χρήσιμες και κακοφόρες συζητήσεις και φυσικά να υποστηρίξουμε την αντιπολίτευση στην διαδικασία αυτή της δύσκολης εισόδου στις διαπραγματεύσεις γιατί για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια έχουμε την κατάπαυση του πυρός η οποία εξακολουθεί είπαμε να κρατεί με σημαντικές βέβαια παραβιάσεις αλλά έχουμε και ανθρωπιστική βοήθεια που παραδίδεται στις πολιορκούμενες περιοχές Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σας παρουσιάσω μια πραγματικά ή ιδιαίτερα ρόδινη εικόνα, αλλά παρόλα αυτά κάποια βήματα επιτέλους ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Ένα από τα βήματα αυτά είναι η μορφή συντονισμού στην οποία αναφέρθηκα πριν για την συντονιστική προσπάθεια της Ρωσίας και της ΙΠΑ ε, σε επίπεδο στρατιωτικό πάντα και ταυτόχρονα η σχεδίαση και η επιβολή της κατάπαυσης του πυρός και η αντιμετώπιση απειλών που θα έφεταν σε κίνδυνο αυτή την εύθραστη εκεχηρία. Αυτοί λοιπόν που μιλάνε για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο πρέπει να ξυπνήσουν γιατί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Τώρα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει και στις δύο task force με διαφορετικό τρόπο και σε σχέση με την κατάπαυση του πυρός σε επίπεδο τασφός είμαστε παρόντες μαζί με άλλες χώρες και οργανώσεις της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης. Είναι παρόντες εκεί και οι συγκεκριτικοί εμπειρογνώμονές μας και δουλεύουμε με τρόπο που θα μας επιτρέψει να συμβάλλουμε στην παρακολούθηση της παύσης των εκδοτασιών μαζί με άλλους φίλους. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ανθρωπιστική βοήθεια, ο ρόλος μας ε, είναι σαφώς μεγαλύτερος, όχι μόνο διότι η Ένωση είναι η καλή, δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές δράσεις, αλλά και διότι στη Συρία συγκεκριμένα ο ρόλος της Ένωσης, και αυτό ήταν πολιτική απόφαση και σωστή νομίζω, δεν ήταν και δεν είναι ενός εμπλεκόμενου επιτόπου. Κάποια κράτη μέλη της Ένωσης είναι, αλλά ο καθοδηγητικός ρόλος εδώ ανήκει στις δύο χώρες που έχουν στρατιωτική δράση και παρουσία και γνώση, αλλά και έλεγχο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν στην διαπραγμάτευση για την πάυση των εχθροπραξιών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μετέχουμε και σε αυτή τη ε, δράση με ενεργή παρουσία εκεί. Και τούτο όπως σας είπα μπορεί να αυξηθεί στο μέλλον. Για την ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής διαδικασίας που πρέπει να ξεκινήσει. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε αναφέρθηκαν πολλοί από εσά στην ανάγκη ενός σχεδίου Μάρσαλ για τη Συρία. Αν δούμε τα νούμερα, τα κονδύλια που δίνουμε στην Συρία, στις γειτονικές χώρες, μπορώ να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το σχέδιο Μάρσαλ με πολύ σημαντικό τρόπο. Η ανθρωπιστική task force όπου όπως είπα παίζει που παίζουμε καθοριστικό ρόλο έχει συναντηθεί τέσσερις φορές, έχει κατορθώσει να μεταφέρει 180 ε, φορτηγά βοήθεια σε 7 πολιοκυμένες περιοχές, βοηθώντας πάνω από 150.000 ε, σύρου σε πόλεις όπω τη Μαντάια, τη Μοντανία, την Αλσάμ, την Κάφνα, την Καφάγια και τον Τερεζόρ. Δεν είναι ένας εξαντλητικός κατάλογος αυτός. Δουλεύουμε αντίθετα για περαιτέρω δράσεις, ούτως ώστε να φτάσουμε σε περισσότερους Σύρους, σε περισσότερες πόλεις της Συρίας σε επόμενες μέρες και εβδομάδες. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε πάνω από 1.700.000 Σύρους μέσα στη Συρία κατά το πρώτο τέταρτο του έτους, τους επόμενους δύο μήνες δηλαδή. Για να βοηθήσουμε απευθείας την ανθρωπιστική παράδοση συνεργαζόμαστε επί τόπου με τους ε, οργανισμούς του ΟΗΕ και γι' αυτό επανενεργοποιήσαμε το γραφείο της ΕΚΟ στη Δαμασκό. Να σας πω, μεταξύ των διεθνών δρόντων η Ένωση είναι η μόνη, πιστέψτε με, που θεωρείται αξιόπιστη από όλες τις πλευρές και εντός Συρίας και στην περιοχή. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια προνομιούχα πρόσβαση σε πολλούς συνομιλητές που πρέπει κατόπιν να προχωρήσουν τα διάφορα βήματα που χρειάζονται για να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στα δύσκολα σημεία. Ο ρόλος μας στην ανθρωπιστική βοήθεια μας επιτρέπει να παίξουμε και σημαντικό πολιτικό ρόλο. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό, να δημιουργήσουμε παράθυρα εμπιστοσύνη με τις διάφορες πλευρές. Ο ρόλος μας είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα αυτά ορθάνυχτα για μια πραγματική, ε, ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση. Πρέπει να έχουμε υπόψη και με αυτά τα θετικά βήματα που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες εβδομάδες ότι μπορεί να υπάρξει νέα κλιμάκωση οποτεδήποτε. Η περιφερειακή κατάσταση είναι έντονη, είναι τεταμένη. Κάθε μέρα μαθαίνουμε ανισχυτικά νέα. Σήμερα το πρωί μία πόλεμος, ε, ένας πόλεμος ενδιαμέσου, ενδιαμέσου, ενδιαμέσου μπορεί πάντα να συμβεί. Εμείς ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια πρόοδος και στο διπλωματικό επίπεδο και στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην προώθηση της κεχηρίας και της παρακολούθησης της κεχηρίας με τον κίνδυνο πάντα όμως να πάμε πίσω αν δεν υπάρξει επαρκής παρακίνηση και επαρκή συνέπεια από όλες τις πλευρές. Αν δεν πιέσουμε Ιδίω και πρωτίστω το καθεστώς, αλλά όλους τους εμπλεκόμενου φορεί να μπουν σε μια πραγματική ουσιαστική πολιτική διαδικασία. Είχα συζητήσεις απευθεία αυτές τις ημέρες με όλους τους εταίρου μας, φίλους, συνομιλητέ, μη φίλους, μέσα στη Συρία, έξω από τη Συρία, για να περάσω το ίδιο μήνυμα, για να προχωρήσουμε στην ανθρωπιστική πολιτική να συνεργαστούμε ούτως ώστε να βελτιωθεί και να κρατήσει η εκεχηρία. Χτες μόλις το συζήτησα με τους Τούρκους εταίρους μας. Αν δείτε το ανακοινοθέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χθες θα δείτε μία μνήα στην ανάγκη συνεργασίας για την βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθήκων σε όλο ένα και περισσότερε περιοχέ μέσα στη Συρία. Αυτό είναι κοινή δέσμευση που συζητήσαμε χθε με του Τούρκου. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρία. Πολύ μικρό. Πρώτα, θέλουμε να μην κλείσει και να, δεύτερο, να ανοίξει περισσότερο. Ανθρωπιστικά, εκεχηρία και πολιτικά. Και με την ίδια ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμπιστούρα για την εξαιρετική συντονιστική δουλειά που κάνει. Οι επαφές μας είναι σε καθημερινή βάση και ο τρόπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΟ σε όλα αυτά τα ζητήματα αποτελεί παράδειγμα και για άλλους τομείς. Νομίζω ότι είδαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει η διπλωματία. Το είδαμε και από πρόσφατες εμπειρίες μας από πέρυσι. Και το Ντάες μπορεί να ιτηθεί, το Ισλαμικό κράτος μπορεί να ιτηθεί. Μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος στην Συρία και να έχουμε και μια διαδικασία μετάβασης στη Δαμασκό. Ξέρουμε ότι μπορούν ε, να ενωθούν οι δυνάμεις στο εσωτερικό της Συρίας για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Και αυτά είναι αποτελέσματα της ιδιαίτερα αποφασιστικής ε, και συνεπούς δουλειάς που έχουμε κάνει. Μετά από πέντε χρόνια τέτοια σκληρής δουλειάς, η διπλωματία, η ευρωπαϊκή διπλωματία, αρχίζει τώρα να αποδίδει κάποια αποτελέσματα. Αλλά οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσαν όλα αυτά να ανατραπούν αν όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν συνεχίσουν με την ίδια σκληρή δουλειά και την ίδια επιμονή που έχουμε δείξει κατά τους τελευταίους μήνες. Η Συρία που καταστράφηκε τα τελευταία πέντε χρόνια δεν θα επανέλθει. Όλες οι ομορφιές και ο πλούτος της Συρίας δεν θα επανέλθουν, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε το λαό της Συρίας να επανέλθει, να ενωθεί με την θρησκεία του, τον πολιτισμό του, με τρόπο ενωμένο και όχι διχασμένο με μια κυβέρνηση πολυσυλλεκτική που θα εγγυάται σε όλους τους ήρους την θέση τους στη χώρα χωρίς να δίνει καθόλου χώρο στο Ισλαμικό κράτος σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν της χώρας και με το μέλλον της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Μογκερίνη για την δήλωσή της. Θα ακούσουμε τώρα τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Πρέντα, 1,5 λεπτό από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, χαίρομαι που σας άκουσα να εμένετε στο γεγονός ότι η σύγκρουση έχει πια διάρκεια πέντε ετών, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς περίοδου δεν είχαμε πολλούς λόγους να ελπίζουμε. Συχνά αυτό δεν το βλέπατε στο παρελθόν. Η εκεχηρία που ξεκίνησε από τις 27 Φεβρουαρίου είναι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό στοιχείο και επίσης πολύ σημαντικό και συμφωνώ μαζί σας είναι το ότι επιτρέπει πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κατάσταση απελπιστική. Ξέρω ότι αυτό άλλαξε σε σχέση με το όταν είχατε έρθει στην Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Η εκεχήρια επίσης είναι σημαντική διότι παρέχει ελπίδα ε, που πρέπει να κρατήσουμε για μια πολιτική διέξοδο. Προφανώς δεν είναι τέλεια η κατάπαυση του πυρός, υπάρχουν ακόμα θύματα, αλλά υπάρχει, εν γέννη γίνεται σεβαστή και είναι μια ευκαιρία για να ξεκινήσουμε προς μια αξιόπιστη πολιτική μετάβαση που δεν σημαίνει προφανώς ε, εκλογές τώρα όπως θέλουν προ προτείνει ο Ασάντι ο Πούτιν είναι αυτό απαράδεκτο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενευτική διαδικασία και όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση θα προχωρήσουμε σε εκλογέ. Ευχαριστώ. Μποστινάρου για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Δύο λεπτά. Κυρία Υπατή Εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν Θέλω να συγχαρώ την είπατε εκπρόσωπο που ξεκίνησε αυτή την πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και για τον πολύ σημαντικό τρόπο με τον οποίο συντονίζει εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους περιφερειακούς ε, φορείς για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή την σύραξη που συνεχίζεται επί χρόνια. Οι τελευταίες δέκα μέρες ήταν οι πιο ήσυχες μέρες για τους περισσότερους Σύρους, οι πιο ήσυχες μέρες που έχουν ζήσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα μπορούσαν αυτές οι μέρες να βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια δυναμική πίσω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες σε αυτή τη χώρα που σπαράσεται από τον πόλεμο ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν και οι ειρηνευτικέ συνομιλίε σύντομα. Μόνο μια πολιτική λύση ε, μπορεί ε, να βοηθήσει και χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική δέσμευση για να το επιτύχουμε. Μια πολιτική λύση στη Συρία θα επιτρέψει τη διεθνή κοινότητα να επικεντρωθεί στα πιο σημαντικά στοιχεία, την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτου και όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων και να τι εμποδίσει να εξαπλωθούν και να ε, εξαπλώνουν τον πόλεμο σε όλη την περιφέρεια θα επιτρέψει στη Συρία, στους, στους Σύρους της Συρίας να παραμένουν στα σπίτια τους και να μην διακινδυνεύουν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη ή αλλού. Η συμμετοχή της μετριοπαθούς Συριακής Αντιπολίτευσης στις διεθνείς συνομιλίες είναι ε, ουσιαστική και πρέπει να είναι εγγυημένη και επομένως ε, καταγγέλουμε κάθε δράση εναντίον των μετριοπαθών ε, Σύρων της Αντιπολίτευσης και εναντίον της πόλης του Χαλεπίου που είναι κατά των διεθνών συνομιλιών. Πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι αυτονόητο ότι η ανθρωπιστική κρίση θα συνεχιστεί αν οι συνομιλίες δεν αποδώσουν καρπούς πολύ συχνά υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φορείς ε, στη σύραξη αυτή στη Συρία. Θα πρέπει όλοι, συμπεριλαμβανομένοι τη Τουρκία και τη Ρωσία, να παραμείνουν στα συμπεράσματα του ψηφίσματο 224, ούτω ώστε να μπορεί να βρεθεί μία λύση για τη Συρία. Ευχαριστώ. Κύριο Τάνοκ, ένα λεπτό για την ομάδα του ECR. Η εύθραστη εκεχηρία στη Συρία προσφέρει στη διεθνή κοινότητα την πολιτική ευκαιρία να πιέσει για την εφαρμογή της αρχικής ειρηνευτικής συμφωνίας της Γενέβης. Έχει σημασία να υπάρξει μια διαρκής ρύθμιση ε, η οποία θα έχει μια κυβέρνηση, θα προβλέπει, θα περιλαμβάνει μια κυβέρνηση στη Δαμασκό που να εκπροσωπεί το σύνολο των Σύρων και να σταματήσουν και αυτοί οι κατανάθεση πόλεμοι οι οποίοι φέρνουν σε σύγκρουση και ε, διάφορες ομάδες ακραίων ε, όπως επίσης και εκπροσώπους της Ίσης στην Συρία. Θα πρέπει επίσης να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των ε, μετριοπαθών ομάδων αντιπολίτευσης για να αποτραπεί μια περαιτέρω έξοδος προσφύγων ε, κάτι το οποίο θα λειτουργήσει εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις βάρος της πολιτικής της κυρίας Μέρκελ. Η πολιτική της Ρωσίας θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να καταστεί ένας αξιόπιστος ε, ε, πολιτικός συνομιλητής. Σα και δύο λεπτά εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Κάθε προσπάθεια για να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία μέσω διαπραγματεύσεων πρέπει να υποστηριχθεί. Αλλά η αδίποτε διέξοδος δεν μπορεί να είναι η λύση. Το πρώτο βήμα είναι να υπάρξει η εκεχηρία, η κατάπαυση του πυρός μάλλον. Έχουμε δει να προκαλούνται για πάρα πολλά χρόνια τεράστιες τραγωδίες απαιτείται να στηρίξουμε τους Σύρους περαιτέρω και θα πρέπει να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική μας θέση. Να αναπτύξουμε μια ενιαία και σοβαρή πολιτική, αν το είχαμε κάνει στο παρελθόν, τότε θα είχαμε αντιμετωπίσει καλύτερα. Τώρα πληρώνουμε τις συνέπειες της αδράνειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει προς τα έξω την μεγάλη της αδυναμία κυρίως να προσφέρει καταφύγιο σε αυτούς που το χρειάζονται. Είμαστε κομβικός παίκτη στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να σταματήσουμε την πηγή της τραγωδίας. Η Ρωσία εξακολουθεί να ενισχύει τον Ασάντ και διαπραγματεύεται ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Πούτιν λειτουργεί ασκώντας την κοινική βία βομβαρδισμού των αμάχων και των νοσοκομείων με, με το άλοθη ότι καταπολεμά τον Τέτοιου είδους συμπεριφορές από την Ρωσία του Πούτιν πρέπει να προκαλέσουν κυρώσεις και θα θέλαμε νέα μέτρα και αντίμετρα εις βάρος της Ρωσίας. Άκουσα ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων δεν θα ξεκινήσει αύριο αλλά τη Δευτέρα η παρακολούθηση της συμφωνίας αυτής γίνεται ξαφνικά κάτι το ακόμα πιο σημαντικό όπως και η παρακολούθηση της, ε, ε, της ε, βοήθειας η οποία δίδεται. Πώς το οργανώνεται αυτό. Αναφερθήκατε στα πακέτα για το Λίβανο και την Ιορδανία. Αρκεί αυτό ανησυχώ πολύ για τον Λίβανο ε, δίνουμε την προσοχή μας και δίνουμε βάρος στην Τουρκία αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε να καταρρεύσει ο Λίβανος. Και επίσης πώς ε, χρησιμοποιείται σαν μοχλό επιρροή στις επαφές ε, με την κυβέρνηση στην Τεχεράνη για να υπάρξει επιτέλους ένα τέλος στο βίο καθεστώς του Ασάντα. Η κυρία Ματίας εξ ονόματος της Γκουε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Μογκερίνη για τις ε, διευκρινήσεις σας. Όντως ε, βρισκόμαστε σε μια φάση εκεχηρίας. πολύ ευάλωτης και πολύ σύνθετης. Ε, είδαμε ωστόσο ότι υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, που θέτει και άλλους όρους, όρους όπως τον αποκλεισμό ενός βασικού ή της Τουρκίας που ζητούν τον αποκλεισμό βασικών παραμέτρων παραγόντων όπως είναι οι Κούρδοι της Συρίας. Θέλω να αμφισβητήσω την θέση του κυρίου Ποστούρα ο κύριος Δημιστούδα είπε ότι η λύση πρέπει να είναι συριακή λύση και ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να εξαρτηθεί από τον συριακό λαό. Θα ήθελα να ξέρω πότε θα έχουμε εμείς μια αυτόνομη θέση που θα εξαρτάται από την θέση των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας ή των υπόλοιπων πλευρών. Μια λύση που θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον Συριακό λαό, που θα πρέπει να αποφασίσει μόνος του το μέλλον του. Για 1,5 λεπτό Κυρία Λόχπιλντερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία και χειρίας ισχύει στη Συρία, αλλά είναι πολύ ευάλωτη και οι συνομιλίες στην Διενέβη ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε ε, να λάβουν χώρα. είναι πολύ σημαντικό για τη διαδικασία των ε, ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων να συμπεριλαμβάνουν όλες ε, τις ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των Κούρδων οι γυναίκες από την πλευρά και της ε, αντιπολίτευσης ε, παίζουν σημαντικό ρόλο και ε, δεν θα πρέπει να μένουν στο περιθώριο. Σήμερα λοιπόν που είναι και η Διεθνής ημέρα της γυναίκας θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα σε αυτές τις γυναίκες στις, και στο καθεστώς του Ασάντ και στην αντιπολίτευση αυτές ε, ε, οι γυναίκες είναι αντικείμενο μιας ταινία ε, των γυναικών που στο Χαλέπι δουλεύουν είτε σε υγειονομικές υπηρεσίες είτε παρέχουν βοήθεια σε άλλες γυναίκες και θα ήθελα να τονίσουμε το ρόλο αυτών των γυναικών που έχουν ε, πληρώσει και με τη ζωή τους όπως ε, η Λουκία Χασέρα είναι μια Κούρδα που είχε ε, δημιουργήσει ένα δικό της blog και δολοφονήθηκε. Ελπίζω ότι στην ενευτική διαδικασία θα προωθηθεί ο ρόλος των γυναικών και από τα Ηνωμένα Έθνη ούτως ώστε να μπορούν να έχουν λέγην στην ενευτική διαδικασία. τα εγκλήματα τα οποία ε, συμβαίνουν στη Συρία κατά των γυναικών και των παιδιών θα πρέπει να καταδικαστούν και θα πρέπει για να υπάρξει μια διαρκή ειρήνη οι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα να τιμωρηθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καστάλντο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι. Βλέπουμε ένα δηλώ βήμα προς τα εμπρός. Στέκει η ανακοχή, μπαίνουν και άλλες ε, ομάδες της διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, το κλίμα βελτιώνεται και από τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία και από τη νίκη των μεταρρυθμιστών στο Ιράν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μη συνεργασία άλλων συμμάχων αυτών των, δύο πλευρών, ιδίω της Τουρκίας και της Οδικής Αραβίας η ημερήσια διάταξη της Τουρκίας δεν ευθυγραμμίζεται καθόλου με την εξωτερική μας πολιτική με δεδομένο το στόχο της να έχει πλήρη και από και άμεσο έλεγχο του Συριακού Κουρδιστάν και των βομβαρδισμών προς τους ε, Κούρδους που χτυπούν και αγωνίζονται κατά του Ντάες. Λίγες προσπάθειες έγιναν επίσης να καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση πετρελαίου που χρηματοδοτεί εμπολή στον ΤΑΕΣ. Η αποδοχή από πλευράς μας όλων των τουρκικών όρων και παραχωρήσεων δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ως ένα μήνυμα αδυναμίας μας με το οποίο στην ουσία προσπαθούμε να πληρώσουμε την Τουρκία για την προσφυγική κρίση αγνοώντας αυτό που γίνεται στην νοτιοανατολική Τουρκία και στο Συριακό Κουρδιστάν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τα δύο πακέτα που αναφέρατε προηγουμένω για τον Λίβανο και την Ιορδανία που καταβάλουν τεράστιε προσπάθειε. Ο δε ρόλο τη Ένωση πρέπει να είναι καθοριστικό όχι μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια και το μέλλον τη ανοικοδόμηση, αλλά και για ένα οδικό χάρτη οριστικού χαρακτήρα η πολιτική επίλυση. Η κύριε τέτοι μα λοιπόν πρέπει να είναι μέρη, μέρη, μέρη τη λύση και όχι μέρη του προβλήματο. Ευχαριστώ. Σαφχάουζερ, ένα λεπτό για το ENF. Δύο παρατηρήσεις, Επίτροπε. Η πρώτη αφορά την Τουρκία. Έχουμε μια χώρα αντιδημοκρατική, το είδαμε τα τελευταία γεγονότα, που υποστηρίζει τον Ισλαμισμό, το αναγνωρίζουν όλοι, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στο Ιράκ και στη Συρία μια χώρα η οποία υποστηρίζει και το οργανωμένο έγκλημα και όμως θέλετε η Ευρώπη να υποκύψει μπροστά στην Τουρκία προστατεύοντας ίσως τα συμφέροντα μιας Ευρώπης ή τα συμφέροντα μιας καγκελαρίου που πρόδωσε το λαό της, που πρόδωσε την Ευρώπη από μια χώρα που δεν ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά κριτήρια. Είναι φυσικό κάτι τέτοιο. Δεν θέλετε να διαλύσετε έτσι την Ευρώπη μέσω των χωρών που θα εξεγερθούν. Δεύτερον, ο μοραλισμός σας ε, συνετρίβει στη σύγκρουσή του με την πραγματικότητα. Εσείς υποστηρίξατε το να υποκύψετε απέναντι στα αφεντικά στους Ηνωμένου Πολιτείε, στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία, στην, στον εκβιασμό. Είναι σαφές λοιπόν ότι εμείς εδώ θα παίξουμε ένα ρόλο βοηθητικό. Αυτό τον ρόλο πληρώνουν όσοι αγνοούν την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόρβιν Μίκε, μη εγγεγραμμένο σε ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη. Επιτρέψτε μου να σας πω λίγα λόγια αλήθειας. Οι ρωσικές εμπλοκές στην Συρία δυστυχώς δεν θα οδηγήσουν στην αποχώρηση της Συρίας. και δεν θα μας επιτρέψει η Ρωσία να απομακρύνουμε τους δικτάτορες. Βέβαια σε περιοχές όπως η Συρία μόνο οι δικτάτορες μπορεί να προστατεύσουν κάποιες μειονότητες από ό,τι φαίνεται όπως οι Δρούσοι και άλλες μειονότητες. Αν προσπαθήσετε να επιβάλλετε τη δημοκρατία στην περιοχή αυτή ε, προφανώς θα αποτύχετε. Όταν μίλησα σε Κούρδους τους είπα ότι θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τον Ασάντ. Μίλησα και με τον Ασάντ και του είπα ότι πρέπει να συμβιβαστεί με τους Κούρδους και συμβαίνει σιγά σιγά αυτό παρά τις αρχικές δια, διαθέσεις τους και δεν θα πρέπει οι διεφθαρμένοι Τούρκοι να καταστρέψουν αυτή την εύθραστη συμφωνία. Ακούσαμε τις πολιτικές αθλητικέ ομάδε, τώρα γενική συζήτηση. Κύριε Γκάμπριελ, ένα λεπτό. Η κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία ε, είπατε εκπρόσωπε. Συμφωνούμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα με την ανθρωπιστική βοήθεια και τι προσπάθειε συνομιλιών ε, στη Συρία, αλλά παραμένει έθραυστη η κατάσταση, όπω είπατε, και γι' αυτό χρειάζεται κάθε μα ε, προσπάθεια. Ε, σήμερα, την Διεθνή ημέρα τη γυναίκα, ο ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στέφαν Τιμιστούρα, υπενθύμησε ότι οι γυναίκε αποτελούν τμήμα μια βιώσιμη και μόνιμη λύση. Έχουν το δικαίωμα ε, και όχι μόνο το καθήκον να συμμετέχουν σε αυτήν την ειρηνευτική διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι είναι κέρια σημασία ε, ο ενδοσυριακό διάλογο. Δεύτερον, αν το ότι έχουμε μείνει έξω από την εκεχηρία μια και δεν συμμετέχουμε στρατιωτικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να συμμετάσχουμε στον ειρηνευτικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να αποτελέσει μια εξισορροπιστική δύναμη και σας ευχαριστούμε κυρία Ήπατη εκπρόσωπα για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ε, προς ε, ε, την οργάνωση μελλοντικών εκλογών. Πώς να οργανωθεί μια διαδικασία εκλογών με 8 εκατομμύρια εκτοπισμένους. θα πρέπει όλες οι χώρες υποδοχής να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα ερώτημα προς σας από τον κύριο Σάνι. Δέχεστε την ερώτηση. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητέ συνάδελφε, σωστά παρουσιάσατε την κατάσταση, αλλά θα ήθελα με την ερώτησή μου να μπω σε ακόμη μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Πιστεύετε ότι μόνο οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνε, δεν είναι υπεύθυνη και η Ρωσία, διότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί δημιούργησαν περισσότερου πρόσφυγε από ότι ε, στο παρελθόν. Πώς νομίζετε λοιπόν ότι θα μπορούσε να συμμετέχει η Ρωσία στη διαδικασία αυτή. κυρία Γκαμπριέλη. Νομίζω ότι στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να έχουμε κατά νου το μήνυμα το οποίο ακούσαμε από την ύπατη εκπρόσωπο. Προσέξτε, διότι πολύ γρήγορα μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως τις κατηγορίες και τις κρίσεις που εκφέρουμε. Όλοι μαζί, η διεθνής κοινότητα ενωμένη θα πρέπει με την ευθύνη που έχει και με το όραμα που έχει να μπορέσει να επαναφέρει τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κύριος Χάουιτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν συζητούσαμε το θέμα της Συρίας ε, στο Κοινοβούλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα επικρατεί απογοήτευση και την περασμένη εβδομάδα ακόμη δεν ε, ελπίζαμε ότι θα μπορέσει να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Ευτυχώ, οι σκεπτικιστές ε, απεδείχθηκε ότι είχαν άδικο και ε, σύμφωνα με ε, δημοσιεύματα σήμερα το πρωί είδα ότι για αρκετέ ημέρε υπάρχει και χειρία και κατάπαυση του πυρό και έφτασαν αποστολέ ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία η ύπατη εκπρόσωπο θα πρέπει να έχει την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να, προχωρήσουμε ούτω ώστε η προσωρινή εκεχηρία να μετατραπεί σε διαρκή ειρήνη. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους και από όλους εκείνους που υποφέρουν στη Συρία γιατί θέλω να μιλήσω και για αυτούς τους συμπατριώτες μου που προσπαθούν ε, το τραγικό θέμα των προσφύγων από τη Συρία να το χρησιμοποιήσουν για τη συζήτηση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για το κατά πόσο θα παραμείνει η Βρετανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο Μπόρις Τζόνσον παραδείγματο χάρη που επαναλαμβάνει τον ε, πλαστό μύθο ότι είναι οικονομικοί μετανάστες αυτοί που έρχονται ως πρόσφυγες από τη Συρία ή αυτό που λέει ο ηγέτης του UKIP που μιλάει για τζιχαντιστές που έρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και ε, ισχυρίζεται ότι θέλει να αποφύγει τους σχετικούς κινδύνους. Είναι ε, επονίδιστοι αυτοί οι άνθρωποι διότι ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς θέλουμε να επιλύσουμε την κρίση αυτών των προσφύγων και οι επονίδιστοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κερδίσουν. Η χώρα μας θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί μια χώρα από μόνη της, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να συνεισφέρει στην ε, ειρήνη ε, στην ε, Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ερώτημα προς εσάς κύριε Χάουιτ. Από τον συνάδελφο Νούταλα. Μπορεί να ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς ο κύριος Χάουιτ διαφωνεί με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τίμεμανς, που είπε ότι οι πλειονότης όσων έρχονται στην Ευρώπη δεν είναι από τη Συρία. Διαφωνεί με τα επίσημα στοιχεία σύλλου στη Βρετανία που λένε ότι η πλειοψηφία όσων ήρθαν στη Βρετανία για άσυλο ήρθαν από την Ερυθρέα, όχι τη Συρία. Μα ε, μας φομίζετε κύριε Χάουιτ, παίζετε ένα πολιτικό παιχνίδι. Απαντήστε λοιπόν διαφωνείτε με τα επίσημα στοιχεία της ε, Βρετανικής Υπηρεσίας Ασύλου. Κύριε Χάουιτ, απάντηση. Είτε και η Κομισιόν και η Πατερμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες αναφέρουν ότι η κύρια χώρα προέλευσης της πλειοψηφίας των προσφύγων είναι η Συρία και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πραγματικοί πρόσφυγες που διώκονται και είναι θύματα ενός εξαετούς εμφυλίου πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει στη διεθνή διπλωματία για να ε, επιτύχει την ειρήνη. Απορρίπτουμε τις, ε, τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Ο κύριος Φώτιγκερ για ένα λεπτό. κυρία Ευχαριστώ πολύ. Μία επιμέρους κατάπαυση του πυρός είναι αυτό το οποίο κατάλαβα σαν πιο σωστό από ό,τι ακούσαμε και σε σχέση με τους συμμετέχοντες και σε σχέση με τη γεωγραφική κάλυψη. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω εδώ ένα αποτελέσματα στα οποία έχουμε καταλήξει είναι η ενίσχυση του ρόλου του Ασάντα και η επανεγκατάσταση της Ρωσίας στην διεθνή σκηνή. Η κατάσταση ως έχει σήμερα επιτρέπει το Ιράν να επανέλθει στην περιοχή. Ίσως κάποιες άλλες συνέπειες να μην είναι τόσο σαφείς όπως αυτές που προανέφερα. Δυστυχώς το ΝΤΑΕΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί και εκτός συνόρων του Ιράκ και της Συρίας. Και οι φρικαλαιότητες δυστυχώς θα συνεχιστούν. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση, μπλε κάρτα έχετε για την κυρία Φώτιγκα ο κύριος Φρουτζούλιτσα για την κυρία Φώτιγκα. Αγαπητέ συνάδελφε, αναφερθήκατε στις φρικαλαιότητες οι οποίες έγιναν στη Συρία και φυσικά στο Ιράκ. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προωθήσει την δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για την Συρία και το Ιράκ έτσι ώστε να γνωρίζουν οι ηγέτες του Νταές ότι θα είναι υπόλογοι και θα δικαστούν για τις φρικαλαιότητες τις οποίες έχουν προκαλέσει εις βάρος και τον Γιαζιντή. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ με την άποψή σας. Λοιπόν θα δώσω τώρα το λόγο τον συνάδελφο Αουστρεβίσιους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, συνάδελφε, πέντε χρόνια σύγχυσης, πέντε χρόνια αδράνειας μας οδήγασαν εδώ που είμαστε σήμερα. Και υπάρχει μια κάποια κατάπαυση του πυρός κάτω από ανεξέλεγκτες συνθήκες. Το συριακό παζλ δυστυχώς το μετακινεί συνεχώς ο Πουτίνα εμείς δεν εμποδίσαμε τους μαχητές να πάνε στο Ίσις και δυστυχώς ο Ασάντ συνεχίζει να προκαλεί τεράστιες προσφυγικές ροές, βομβαρδίζει σχολεία και νοσοκομεία και ψευδείς ιστορίες προπαγάνδας. Τώρα θα πρέπει ε, να είμαστε φίλοι μαζί τους. Δυστυχώς στρατιωτική λύση ε, είχε υποθεί μέχρι τώρα δεν μπορεί να υπάρξει στην Σύρια. Ε, πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση, ποιο θα είναι το τίμημα για την λύση αυτή και ποιος θα πληρώσει το συγκεκριμένο τίμημα. Ο κύριος Κούζο Περμούη κατάπαση του πυρός είναι ένα καλό νέο, είναι μια προσπάθεια πολιτική η οποία βέβαια είναι μακράν μιας διαρκούς ειρήνης για τη Συρία. Εμείς υποστηρίζουμε αυτά τα οποία κάνει ο κύριος Ντεμιστούρα αλλά ενθυμούμαστε πριν δύο-τρία χρόνια τις δηλώσεις ε, οι οποίοι έλεγαν τι καλή που ήταν τότε η Αλ δηλαδή η Αλ Κάιντα. Βλέπουμε ότι δυστυχώς όλες αυτές ε, οι ε, ευχές του παρελθόντος δεν οδήγησαν πουθενά. Θα πρέπει να βρούμε ένα ανεξάρτητο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να το κάνουμε αυτό συνεργαζόμενοι με τους συμμάχους μας, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Και φυσικά η τουρκική κυβέρνηση ε, η ίδια παραβιάζει την ανακοχή και φυσικά οι διαπραγματεύσεις δεν συνεχίζονται στη Γενέβη όπως θα θέλαμε. Σμιτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και κυρία Μογγερίνη, ευχαριστώ για μια πολύ εντυπωσιακή ενημέρωση για την κατάσταση στην Συρία. Και εγώ συμφωνώ με το, τους επένους προς τον κύριο Μιστούρα και εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά η Ένωση δεν παράγει και δεν, πουλά, και δεν παράγει όπλα και βόμβες, αλλά δουλεύει για να διευκολύνει ένα διάλογο που οδηγεί σε αποτελέσματα. Η, το κόμμα μου θέλει να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσουμε ως Βρετανία να μετέχουμε σε αυτό το πλαίσιο ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως, αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η σωστή περιγραφή. Η εκεχηρία στέκει. Είναι σημαντική η συνέχιση της βοήθειας προς τον Λίβανο και την Ιορδανία που είναι πολύ ευάλωτες χώρες. Επίσης, λογοδοσία. Πρέπει να υπάρξει λογοδοσία όλων των πλευρών, όλων των παρατάξεων και χαίρο που ανοίξατε στη Δαμασκό γραφείο του ΕΚΟ. Ε, πώς βοηθάτε όμως σε διεθνές και τοπικό επίπεδο ΜΚΟ για να συλλέξετε στοιχεία που θα εξασφαλίσουν ότι, όταν, ε, ότι η λογοδοσία θα είναι στοιχείο της λύσης στην Συρία. Νάταλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όπως γνωρίζουμε, η Συρία είναι ενδεχομένω το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια κοινότητα. Βλέπουμε ε, την φρίκη του Ισλαμικού καθεστώτος, τα, ε, τις τηλεοπτικές απεικονίσεις ε, αποκεφαλισμών, της θανάτωση στην οθόνη και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2013 όλη η δυτική πολιτική και ο Τζον Μακέιν και ο Γκίφερ Χόφστετ από τη δική μας πλευρά μας έλεγαν ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε τους επαναστάτε, μεταξύ των οποίων και την ε, Ανούσρα. ευτυχώς που δεν το κάναμε. Γιατί δεν συνεχίζουμε να κάνουμε τίποτα για την Σαουδική Αραβία και γιατί συνεχίζουμε να δίνουμε χρήματα στην Τουρκία και να καλούμε την Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εκείνη είναι υποστηρικτή τη Τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Όμπερ Μάιερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί με εκταμιεύσεις δισεκατομμυρίων να βοηθήσει την Τουρκία οδηγούμενη σε ένα σφάλμα. Η Τουρκία δεν είναι ε, ευκταίος εταίρος για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ειρηνευτική διαδικασία από καμία πλευρά με τη βοήθεια ε, φιλοτουρκικών στρατιωτικών ομάδων να διεξάγεται πόλεμο στα σύνορα με την Τουρκία και καταπατείται το διεθνές δίκαιο διαδικασίες ε, κατά ε, της Άγκυρας οδήγησαν σε κατάπαυση ε, του πυρός. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε και με το καθεστώς του Ερντογάν δεν μπορούμε με τέτοιο καθεστώς να κάνουμε προόδους στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Μίλιαν Μον, ένα λεπτό. Πρόεδρε, η συμφωνία και η χειρία στη Συρία παρέχει ελπίδες και ελπίζω να ενισχυθεί με τις επόμενες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Είναι αναγκαία η εκεχηρία, δεν είναι πλήρης, αλλά έχει μειωθεί η βία και Προφανώς δεν είναι η λύση στην σύραξη. Πρέπει οι διαπραγματεύσεις που θα προχωρήσουν ξεκινήσουν να δώσουν πολιτική λύση βάσει του ανακοινοθέντου βάσει των όρων του ανακοινοθέντου της Γενέβης του 2012. Η έλλειψη πρόοδου σε πολιτικό επίπεδο ενισχύει την παγίωση δομών όπως το ΤΑΕΣ και τις δυσχέρειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και χαίρο κύριε Μογκερίνη που δεσμευθήκατε με την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων της Γενέβης και, της, ε, ε και του Αραβικού Συμβέσμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Συρίας. Οι διεθνείς ε, δρόντες πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ούτως ώστε να υπάρξει μια λύση τελικά στην σύραξη της Συρία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Δύο λεπτά. Νομίζω ότι ο αγώνας των Σύρων εναντίον του Ασάντα μετετράπη σε εμφύλιο πόλεμο και σε κατανάφεση πόλεμο ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και την Τουρκία καταστρέφοντας τη χώρα και δημιουργώντας πάρα πολλά προβλήματα και μεγάλη δυστυχία εις βάρος ε, των ε, σύρων πολιτών. Η παρέμβαση των Ρώσων δυστυχώς καλύπτει ένα κενό. Τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν με συντονισμένο τρόπο, δεν μπόρεσαν να επιλύσουν την σύραξη μέσω μιας σωστής πολιτικής, προσπαθώντας να καταπολεμήσουν τους τρομοκράτες. E Νομίζω ότι έτσι ε, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τα παιδιά. Υπάρχουν ε, επίσης ε, πάρα πολλοί οι οποίοι προσπαθούν να καταφύγουν στην Ευρώπη είναι άνθρωποι κατεστραμμένοι που θα καταλήξουν τη μία μέρα, μία μέρα στα χέρια των τρομοκρατών. Νομίζω ότι πρόβλημα θα έχουμε και στην Λιβύη όπου η ασφάλειά μας ε, απειλείται. Δεν μπορούμε από μόνοι μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσουμε τη σύγκρουση αλλά πρέπει να συγχαρώ επιτέλους την κυρία Μογκερίνη. Η κυρία Μογκερίνη κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει έτσι ώστε να υπάρξει μια κατάπαυση του ε, πυρός απαιτείται η Ευρώπη να λειτουργήσει αλληλέγγυα, ηγετικά και πρωτοπόρα. Το Συμβούλιο ε, έχει προχωρήσει σε ανήθικες συμφωνίες με τον Ερντογάν και αυτό με κάνει να αμφιβάλλω για την ποιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στην εξουσία. Ο κύριος Μπέλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είπατε στην εισαγωγή σας κυρία Μογκερίνη, αναφερθήκατε μάλλον στους Τούρκους εταίρους σας. Υπήρξαν κάποιες εξελίξεις βέβαια σχετικές με την Τουρκία που με ανησυχούν ιδιαίτερα. Δεν ξέρω πως βλέπετε τον ρόλο της Τουρκίας στις περιφερειακές συγκρούσεις γύρω από την Συρία. Αν δει κανείς, τι συμβαίνει. Ε, τα όπλα πολλές φορές προέρχονται από τουρκικά εδάφη και αναπτύσσονται δυνάμεις εναντίον των Κούρδων από τις ε, τουρκικές ε, δυνάμεις. Νομίζω ότι αυτό είναι μια παράδεκτη κατάσταση. Έχουμε να κάνουμε με Τούρκους τζιχαντιστές και ταυτόχρονα <coughs> ελληνικές αρχές σταμάτησαν και ένα πλοίο εμπορικό γεμάτο όπλα που πήγαινε στο Λίβανο για να εξοπλίσει αυτές τις ε, πολιτικές ομάδες. Βάγγελ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Μογκερίνη, μετά από αρκετά χρόνια βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου η ανθρωπιστική καταστροφή μπορεί εν μέρει να επιληθεί δια της πολιτικής διαδικασίας που θέλουμε να οδηγήσει σε ειρήνη στη Συρία. Η ανθρωπιστική καταστροφή ήταν αποτέλεσμα μιας εσφαλμένης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης ε, εσφαλμένης και από δικής μας πλευράς. Στην σύραξη στη Συρία δεν καταλάβαμε πού οδηγούσε η κλιμάκωση των δράσεων στην Συρία. Έχουμε τρία θετικά σημεία. Εκεχηρία, συντονισμός μεταξύ ε, ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας και τρίτον, διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχουν και η Ρωσία και ο Άσαντ. Είπατε ότι δεν είμαστε σε μια κατάσταση ενός νέου ψυχρού πολέμου. Σύμφωνα όμως με άλλους συναδέλφους που άκουσα που δεν εστίασαν την προσοχή τους στη Συρία αλλά που προσπαθούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τον Πούτιν αυτή τη στιγμή βλέπω ότι μια τέτοια κατάσταση θα ήταν εντελώ περιττή. Ε, ε, και θα μπορούσε να πει κανεί ότι βιώνουμε ένα ψυχρό πόλεμο. Θα έπρεπε στην Ευρώπη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά τον πόλεμο στη Συρία. Θα χρειαστεί μια διαδικασία συμφιλίωση στη Συρία. Ντόνι, έχει το λόγο για δύο λεπτά, Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Είμαι πεσμένο ότι η Αγγελία είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Αλλά εκεί ξεπίδησε μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πέρασαν πέντε δύσκολα χρόνια σύγκρουσης και ανθρωπιστικής κατάστασης ε, ανάγκης. Οπότε τώρα είπαμε ότι επιβάλλεται να γίνει πολύ πιο σημαντική παρέμβαση ανθρωπιστική αλλά επίσης θα πρέπει να ξεκινήσει και ένα πολιτικό προτσές μια διαδρομή ούτως ώστε να δοθεί στη χώρα η ευκαιρία για ένα μέλλον που θα το οικοδομήσουν οι ίδιοι. Θεωρώ ότι ε, έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των να είναι αυθεντικός πρωταγωνιστής. Είναι επομένως ε, δική μας ευθύνη από σε εμάς να δώσουμε μια απόκριση, μια απάντηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Άρα θα πρέπει να τονίσουμε τη βοήθεια των ε, πέντε δις και πολύ περισσότερο το οποίο έχουν δοθεί από εμά ως ε, δωρητές. Θα πρέπει επίσης να χτίσουμε κάποια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων περιφερειακά και τοπικά εις αυτή την σύγκρουση στην ε, Συρία. Απαιτείται η ευρωπαϊκή πολιτική παρουσία. Χρειάζεται εκεί να αποκτήσουμε αξιοπιστία, να ρίξουμε ένα αισθητό ειδικό βάρος. Άρα χρειάζεται να γίνει μια εθνική συμφιλίωση. Θα πρέπει να αναλάβουμε επομένω ε, έναν περιφερειακό ρόλο για να φτάσουν στη συμφιλίωση ακριβώς όπως κάναμε και στην περίπτωση του πυρηνικού προβλήματος με το Ιράν. Με την κρίση των προσφύγων είδαμε ποια είναι η πρόκληση, αλλά θα πρέπει να δώσουμε αυτή την διάσταση στην εξωτερική μας πολιτική. Να ακουστεί η φωνή μας ενιαία και να έχουμε συνέπεια σε αυτή την πολιτική. Αν θέλουμε να διδραματίσουμε αυτόν τον ρόλο θα πρέπει να έχουμε σταθερή πορεία, να μην υπάρχουν επομένω οι διαφωνίες και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η ειρήνη πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει είναι απαραίτητη. Από τον κύριο Μπονάνο έχετε περώτηση. Ε, αποδέχεστε. Ναι. Όχι, λέει ο κύριο Παντζέρη. Λοιπόν, στον επόμενο αγωγητή, Ο κύριο Πιοτρόφσκι. Έχετε ένα λεπτό κύριε. Σα ευχαριστώ. Ο πόλεμος στην Συρία έχει ήδη κρατήσει μία πενταετία. Έχει κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές. Είδαμε να φαίνεται κάποια ακτίδα ελπίδας για συμφιλίωση μέσω του ΟΗΕ να πετύχουμε κάποια σταθεροποίηση στην περιοχή. Είναι το κλειδί η ειρήνευση για την λύση του μεταναστευτικού. Άρα θα πρέπει να μπει ένα φρένο ε, στην θυσία τόσων αμάχων. Έτσι, επίσης θα σταματήσει η ροή των ε, μεταναστών και αυτοί που έχουν έρθει θα επιστρέψουν σπίτι τους. Μιλάμε για 135 που πάρα πολύ πρόσφατα έχασαν ε, ε, τη ζωή τους τώρα και πάνω από 500 επίσης ε, σκοτώθηκαν ε, από τον στρατό. Άρα θα πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές ανθρωπιστικές προσπάθειες. Κύριε Σνάρτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αδράνειά μας στην περίπτωση αυτή προκάλεσε κατάρρευση στη Συρία. Παρατείναμε τον πόλεμο, δεν λύσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν και σήμερα Είμαστε ενώπιον μιας πραγματικότητας που δεν αρέσει σε κανένα μας σε ένα πόλεμο οι πορτογαλιστέ δεν είναι αυτοί που θέλουμε εμείς, αλλά οι πραγματική Από τη μια είναι το καθεστώς του Άσαντ που ταυτόχρονα είναι και ε, εγγύηση για τους λίγους Σουνίτε, για τους Ελαουίτες βεβαίως και για τους χριστιανούς, για την ασφάλειά τους και απέναντι έχουμε τους ε, Ουαχαβίτες του Τζιχάτα Νούσρα που είναι τζιχατιδιστέ, ή, ή τα Χαρασάπ που είναι υποτίθεται σύμμαχοι τη δύση, αλλά είναι το ίδιο και κάτι άλλες οργανώσεις εκεί. Έχουμε απόλυτη ανάγκη να ε, ε, καταφύγουμε σε μια ελευτική διαδικασία και να αναγνωρίσουμε ότι η ρωσική επέμβαση ήταν εκείνη που τελικά προκάλεσε αυτό το γεγονός για να συμφωνήσουμε. Το να είναι κανείς ε, πρωτογενός και αφελός ε, αντιρώσος δεν βοηθάει. Μετά από πέντε χρόνια χρειάστηκε να επέμβουν οι Ρώσοι που ενισχύουν ε, ένα καθεστώς εγκληματικό μεν πλην υπαρκτό που είναι αυτό του Άσαντ. Θα πρέπει η Ευρώπη να δράσει με αποτελεσματικότητα κατά της τρομοκρατίας υπέρ της ειρήνης και στρατηγικά κάτι τέτοιο εμείς δεν το πράττουμε. Ο ε, κύριος Χάν, για δύο λεπτά παρακαλώ. Άψε το μικρόφωνο σας, του λέει ο Πρόεδρος. Δεν το άναψα, το άναψα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, εκατοντάδες σύρων χρησιμοποιούν αυτήν την ανακοχή ούτως ώστε να διαμαρτυρούν κατά της κυβέρνησης και καλούν στην ανατροπή του Άσαντ και να υπάρξει μια ενωμένη και ελεύθερη Συρία. Αυτό μας θυμίζει το πώς ξεκίνησαν την άνοιξη του 11 εχθροπραξίες. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιους απόσχηση, Απλώς θα περισταλούν κάπως ε, οι μάχες. Και έχουν ε, σκοτωθεί πάρα πολλοί άμαχοι, άρα θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να μπορέσουμε τώρα να πάμε σε ένα περιβάλλον που θα βοηθήσει διαπραγματεύσει μεταξύ των σύρων. Θα πρέπει αυτές οι διαπραγματεύσει να αρχίσουν να συνεχιστούν και να έχουμε μια γενική κατάπαυση πυρός και να έχουμε και έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό και θα πρέπει επίσης οι Σύροι να έχουν το πιδάλιο, αυτοί θα πρέπει να βρουν την λύση. Οι δε διεθνεί κοινότητε, θα πρέπει καλοπίστως να εφαρμόσει την συμφωνία ακριβώς στη συνέχεια της συμφωνίας του Μονάχου. Επίσης και το Ιράν θα πρέπει να ασκήσει θετική επιρροή και οι άλλες χώρες για να γίνει σεβαστή αυτή η ανακοχή και επομένως θα πρέπει να γίνει προσπάθεια και πολιτικά και διπλωματικά και επίσης να δοθεί βοήθεια παντού στη Συρία. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει φραγμός στην ανθρωπιστική βοήθεια και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση των δωρητών εκεί, οπότε θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να δείξει τόλμη, δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Φέτο να είναι η χρονιά που θα σταματήσει η αιματοχυσία. Είναι κοινό μα στόχο να νικήσουμε το Ισλαμικό κράτο και να δώσουμε τέλο σε αυτή την κρίση. Επομένω, να βοηθήσουμε στην ευκαιρία διαδικασία είναι προ το συμφέρον μα και έτσι να πάμε σε μια κυβέρνηση ε, όλων των ε, σύρων που να είναι βιώσιμοι. Έχετε μία περώτηση, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπουράν θέλει να σας την υποβάλει. Την αποδέχεστε κύριε Καν. Όχι, ευχαριστώ. Καλώς, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα προχωρούμε. Έχουμε τον κύριο Σκρίπεκ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κυρία είπατε εκπρόσωποι, είναι η στιγμή που πρέπει να ειρηνεύσει η Συρία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μία μια ομάδα που θα εκπροσωπεί και τους ασυροχαλδαίους θα πρέπει να προσθεθεί ε, στην ε, ομάδα της Συρίας στις ε, συνομιλίες ειρήνευσης. Πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές έχω ζητήσει να έχουμε αυτοδιαχείριση δημοκρατική στη βόρειο-ανατολική Συρία, γιατί δεν απειλούνται μόνο από το Ισλαμικό κράτος, αλλά και από άλλους. Θα πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει αυτή την περιοχή η Τουρκία. Διαφορετικά θα δούμε κύματα ε, μεταναστών και προσφύγων να πλημμυρίζουν τις γειτονικές χώρες και την Ευρώπη. Θα πρέπει η περιφερειακή κυβέρνηση, η κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση στο Ιράκ να ανοίξει όλες τις, ε, όλα τα περάσματα στο Φισκαμπούρ έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθόλου περιορισμοί. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους γιατί είναι το κλειδί για τη σταθερότητα στην περιοχή. Ε, Υπάρχει ερώτηση για σας κύριε Σκρίπεκ. Την αποδέχεστε. Μάλιστα λέει ο κύριος Σκρίπερ. Καλώς επομένως. Μπορείτε να βάλετε την ερώτηση, την επερώτηση. Ποιος. Ποιος την υποβάλλει. Στέτινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σίτινα, ήθελα να λάβω το λόγο. Στη διαδικασία Κατσιάη ε, δεν ήταν μπλε κάρτα, γι' αυτό σήκωσα το χέρι μου. Ζητώ συγγνώμη, παρεξήγηση για μετά ήτανε. Ο κύριος Πάσκου, για ένα λεπτό. Ε, ε, πρόεδρε, κυρία Υπάτη, εκπρόσωπε, ο εμφύλιος πόλεμο στη Συρία έχει πολλέ επιπτώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγική κρίση, τρομοκρατία, αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση στην περιφέρεια, περίπλοκες σχέσεις με την ε, Συρία, ενδεχόμενη κλιμάκωση. Δύο πρόσφατες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός δεν κατάφεραν να επιφέρουν και χειρία ανάμεσα στο καθεστώς και την αντιπολίτευση και τις διάφορες εκεί φατρίες. Για, κατά κύριο λόγο, επειδή δεν συμφωνούν οι επεμβαίνουσες δυνάμεις περιφερειακές και εκτός περιφέρειας για το μέλλον και τη μοίρα του καθεστώτος Άσαντ και το πώς υποστηρίζει ο καθένα σε πλευρέ. πλευρές θα πρέπει να είναι αποκλειστικά πολιτική η λύση μετά από γνήσια και χειρία και ανθρωπιστική επέμβαση για να βοηθηθεί ο πληθυσμός ο άμαχος που είναι όμοιρος. Θα πρέπει να περάσουμε από ε, το στρατιωτικό στο πολιτικό και στο ανθρωπιστικό σκέλος για να λυθεί αυτή η σημαντική σύραξη στο κατόφλι μας. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο κύριος Λίτς για ένα λεπτό παρακαλώ έχετε το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρία Επάτη εκπρόσωπε. Είμαι υπέρ ε, ε της εκεχηρίας που ε, έχουν οι ε, γενικές γραμμές. Το επόμενο βήμα είναι να επανεληφθούν οι συνομιλίες της Γενέβης για να θέσουν τα θεμέλια μιας βιώσιμης ειρήνης. Μέχρι τότε θα πρέπει όμως να επέμβει το ε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να τιμωρήσει τα εγκλήματα πολέμου. Καλωσορίζω τις πρωτοβουλίε όπως είναι η Επιτροπή για τη Διεθνή Δικαιοσύνη και Λογοδοσία. Την υποστηρίζει και η Γερμανία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι υπάλληλοι εκεί συλλέγουν ε, τεκμηρίωση και υλικό για τον εφήλιο πόλεμο. Έχουν αρκετά πιστήρια και αποδείξει για να μπορέσει να προσαχθεί ενώπιον του Διεθνού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα ο Άσαντ. Το θέμα είναι όμω ποιο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο. Χρειάζεται σύσταση νέου δικαστηρίου. Θα πρέπει όλοι και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία να τα λάβουν αυτά υπόψη. Γενικότερα, το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο της εργαλειοθή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι υπάρχει τμήμα και, υψηλό ε, για τους δικτάτορες που παραβιάζουν ε, τα δικαιώματα των λαών τους. Και συστηματικά θα πρέπει αυτοί να προσάγονται στο, ειδικό, μάλλον στο ποινικό δικαστήριο. Ε, έχετε κάποια ερώτηση κύριε Λίτση και αν δεν υποβάλλει ο κύριος Μπονάνο. Αποδέχεστε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Μόνο ένα θα λάβει το λόγο αναπολιτική ομάδα λαμβάνοντα υπόψη τι αιτήσει σχετικώ όπω ε, με τη σειρά που υπευλήθησαν. Κύριο Σόγκο, έχει το λόγο. Το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε η χώρα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Όμως δεν φαίνεται στον οριζόντα το πέρας του πολέμου. Δεν βλέπω να είμαστε πιο κοντά στη λύση. Μάλλον απομακρυνόμαστε από την ειρήνη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει ιστορική ανωτερότητα γιατί αυτό θα βοηθούσε κατά κάποιο τρόπο οπότε από πλευράς Ευρώπης τι κάνουμε βλέπουμε τα εκατομμύρια που φεύγουν από τη χώρα έρχονται στην Ευρώπη και ξεχνούν την πατρίδα τους δεν έχουν καμία ελπίδα να γυρίσουν οπότε σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε και να τιμήσουμε όλες εκείνες που βοηθούν τις οικογένειες του στη Συρία και στις γύρω χώρες. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τη Συρία θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω ότι υπήρξαν δυνάμεις της Δύσης και φυσικά και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία που στήριξαν τον ΤΑΕΣ. δηλαδή στήριξαν το ακραίο σουνητικό Ισλάμ προκειμένου να χτυπηθούν οι Σιήτες και κυρίως ο Άσαντ και γι' αυτό ενισχύθηκε το Ντάεσ. Αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Η κατάσταση φυσικά στη Συρία είναι κρίσιμη, πρέπει να εντυθεί το Ντάεσ, πρέπει να υπάρξει ειρήνη και χωρίς ειρήνη κυρία Μογκερίνη φυσικά θα συνεχίσουν να έρχονται χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 40.000. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στο τέλος του μηνός θα εγκλωβιστούν 150.000 ε, πρόσφυγες. Εδώ μπαίνει το ερώτημα. Τα Σκόπια και η Αλβανία έχουν κλείσει τα σύνορα ο κύριος μπαν είπε ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. εσείς από την πλευρά σας ως ευρωπαϊκή ένωση ως ύπατη εκπρόσωπος τι θα κάνετε; πρέπει να αναλάβετε ενέργειες για να ανοίξουν τα σύνορα. είναι παράνομο αυτό που γίνεται. δεν μπορεί να εγκλωβίζονται χιλιάδες πρόσφυγες στην ελλάδα. δεν μπορεί η ελλάδα να έχει μετατραπεί σε ένα προσφυγικό νταχάου. ευχαριστώ. Έχετε ένα λεπτό κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόκειται για μια ανακοχή. Αυτό είδαμε ότι προσπάθησαν να πετύχουν σήμερα. Εντάξει η κατάσταση αυτή είναι καλύτερη από τον πόλεμο, άρα μακάρι να συνεχιστεί. Ε, γι' αυτό και σας λέω ότι θα είναι πάρα πολύ θετικό όλοι να εμπλακούμε σε αυτό και εσείς ε, κυρία ε, Επίση είδαμε ότι είναι πλάκια και η Ρωσία να βρει μια λύση, αλλά δεν πρέπει να απόκειται το μέλλον μα ε, τα χέρια των Ρώσων το, η Συρία ανήκει στους Σύρους και σε κανέναν άλλο άρα είναι ξεκάθαρο ότι ο εχθρός είναι το Ισλαμικό κράτος έδειξαν οι τρομοκράτες πόσο εύκολα διαπράττουν φρικαλαιότητες άρα θα πρέπει πάσα απόφαση να ληφθεί από τους Σύρους. Εάν θέλουμε να στήσουμε ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο ε, για τα εγκλήματα πολέμου και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά έτσι κι άλλιω θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις οι Σύροι. Κύριος Επιτίδιος, ένα λεπτό. Grazie, signore Presidente η κατάβαση του πυρός στη συρία είναι το πρώτο ενθαρρυντικό μήνυμα από την εποχή που άρχισε ο πόλεμος στη χώρα αυτή ότι υπάρχει μια ελπίδα να εξομαλυνθεί η κατάσταση σε αυτή την πολύπαθη περιοχή. Ε, ήδη σύμφωνα με πληροφορίες έχουν μειωθεί κατά 90% οι απώλειες των αμάχων και κατά 80% οι απώλειες των εμπολέμων. Εκείνο το οποίο δημιουργεί προβληματισμό είναι η απροθυμία της Συριακής Αντιπολιτεύσεως να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενέβη σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ένωση παρά το γεγονό ότι αυτή συμμετέχει ενεργά τόσο στην παροχή ανθρωπιστική βοήθεια όσο και στην κατάπαυση του πυρό εντούτοις έχει απολέσει μια σημαντική ευκαιρία να αποτελέσει ένα ε, σπουδαίο και σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια σκακέρα διότι α είμαστε ειλικρινεί εάν δεν παρενέβαινε στρατιωτικά η ρωσία η συρία θα είχε καταληφθεί από τις δυνάμεις του isis και θα είχε μεταβληθεί σε μια ακόμη ισλαμική χώρα η οποία θα ήταν εχθρική προς τη δύση και επικίνδυνη για τα συμφέροντά της στην ευαίσθητη περιοχή της ε, μέσης ανατολής. Ehm, Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μπονάνα, στο Καζιά δεν προβλέπετε ερώτηση. Τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πάρα πολύ καλό θα ήταν εάν αυτή η πρόσφατη ανακοχή θα μπορούσε να είναι το τέλος αυτού του πεντήτους πολέμου. Όμως είναι πάρα πολύ ευάλωτη η σαθρή. Έχουμε, είδατε και κάποιο είδους συμμαχία ε, των γερακιών ούτως ώστε να υπάρξει επίθεση κατά των Ρώσων ε, συγκεντρώνονται όλο και περισσότερα όπλα στην ε, περιοχή. Άρα βλέπουμε πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Ε, θα πρέπει να υπάρξει κάποια συμμαχία μεταξύ Ρώσων, Ιρανών, κυβέρνησης, Χεσμπολάχ και έτσι να υπάρξει μια τέτοια συμμαχία ε, και διάφορες άλλες ομάδες ε, έχουν προσκληθεί σε αυτό το μέτωπο από τις ε, ΗΠΑ. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που έρχονται κάθε μέρα στην Ευρώπη. Βλέπουμε πόσο κάθε μέρα μαυρώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν θα πρέπει να αναμειχθούμε με τρόπο που να αποσταθεροποιήσουμε τη χώρα όπως το κάνανε άλλοι. Γιατί όλα θα πηγαίνουν το καλοκαίρι, ήταν ντροπή και βλέπουμε ότι τελικά το σωστό είναι να καθορίσουν το μέλλον τους και να λάβουν τις στήριξη στο χέρι τους οι Σύριοι οι ίδιοι. Ένα λεπτό τελευταίος. Ευχαριστώ Κυρία Πάτη, εκπρόσωπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημαντική σας ε, παρουσίαση αλλά και την σημαντική σας παρουσία στις ειρηνευτικές ε, διαπραγματεύσεις και τη βελτίωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά εδώ ακριβώς δεν αρκεί καθόλου αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικρατεί πείνα ε, στους καταβλισμούς των προσφύγων. Οι άνθρωποι δεν προστατεύονται από το ψύχος αρκετά. Και όσο ισχύει κάτι τέτοιο χρειάζεται να δαπανούμε περισσότερα χρήματα και Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να δώσουμε χρήματα στην Τουρκία για να χτίσει φράχτη και τείχος για να προστατεύεται από τους πρόσφυγες. Δεν έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα να δώσουμε τα χρήματα στους καταβλισμούς για να μην έχει ο κόσμος αιτία να φεύγει, να μπορεί να επιβιώνει στους καταβλισμούς. Σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ να φροντίσετε ε, τουλάχιστον ε, οι στοιχειώδεις ανάγκες ε, του κόσμου να καλύπτονται και να ικανοποιούνται επιτόπου στους καταβλισμούς εκεί. Ευχαριστώ. Για να απαντήσει τώρα, το λόγο έχει η κυρία Μορκερίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας με κάθε ειλικρίνεια πως μερικές φορές μου δημιουργείται η εντύπωση πως είναι σχετικά εύκολο να κάθεται κανείς εδώ και να τονίζει όλες τις ελλείψεις σε μια κατάσταση η οποία εγώ ίδια θα παραδεχθώ απέχει πάρα μα πάρα πολύ από το να είναι τέλεια. Δηλαδή, να παραπονηθώ πως αυτό το ποτήρι είναι μισογεμάτο, μα δεν είναι καν κοντά στο να είναι μισογεμάτο. Όμως πριν μια εβδομάδα ήταν άδειο. Οπότε το δικό μας καθήκον είναι σταγόνα σταγόνα να χτίσουμε και να γεμίσουμε ένα ποτήρι το οποίο κάθε μέρα θα γεμίζει λιγάκι. Γιατί κάθε σταγόνα είναι μια ζωή που σώζουμε και κάθε ζωή που σώζουμε έχει τη δική της αξία είτε στην Ευρώπη, είτε στο Αιγαίο, είτε στη Συρία, είτε στην Ιορδανία ή στο Λίβανο. Η δική μου δουλειά λοιπόν, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας, αλλά η δική μου δουλειά δεν είναι να έρθω εδώ και να σας πείσω με τα επιχειρήματά μου ότι τα πάντα είναι τέλεια. Όχι, η δική μου δουλειά είναι κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε με ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε ως διεθνής κοινότητα η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί ενωμένη γιατί πέντε χρόνια πολέμου είναι το αποτέλεσμα πέντε ετών διεθνούς διέρεσης. Είχαμε σειράξει στη Συρία, γύρω από τη Συρία κοντά στη Συρία. Πιστεύω πως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν είναι αυτός να προσπαθήσει και όπως είπατε πολλοί από εσά, να γεφυρώσει τα διάφορα συμφέροντα. Γιατί έχουμε τόσους παίκτες μέσα στη Συρία και έξω από τη Συρία που έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους που θα διαφωνήσουν για σχεδόν τα πάντα. Όμως επειδή τα δικά μας ζωτικά συμφέροντα, τα πολιτικά και θα έλεγα και ηθικά και τα συμφέροντά μας ως Ευρωπαίοι για θέματα ασφάλειας. Γιατί όσο ε, πιο πολλοί πρόσφυγες πεθαίνουν, τόσο πιο πολύ κερδίζει ε, το Ισλαμικό κράτος και ξέρω πως θα έρθει και ο κύριος μας για να σας εξηγήσει τι γίνεται. Τα δικά μας συμφέροντα λοιπόν για τη διαχείριση των ροών είναι καταρχήν ανθρωπιστικά, είναι κατά δεύτερον πολιτικά και θα πρέπει να εντοπίσουμε ποιος είναι ο κοινός τόπος που θα συγκεράζει πολύ διαφορετικά συμφέροντα έτσι ώστε βήμα-βήμα να διευρύνουμε τον κοινό αυτό τόπο που θα επιτρέψει στη διεθνή κοινότητα και τους περιφερειακούς παίκτες να διευκολύνουν και όχι να καταστήσουν αδύνατον για τους Σύριους να ζουν μαζί και όχι να ε, είναι σε εμφύλιο όπως γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν μπορούμε καν να τα πούμε ανακοχή. Όχι, μιλάμε για διακοπή εχθροπραξιών. Καταλαβαίνετε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα. Άρα λοιπόν ακόμα γίνεται πόλεμος. Δεν θα εξεφανιστεί ο πόλεμος αυτός την επόμενη εβδομάδα. Και το είπα στην αρχή ξεκάθαρα και μπορεί να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση όπου επιτόπου η κατάσταση θα χειροτερεύσει γιατί δεν έχουμε καταφέρει να προωθήσουμε όλα αυτά τα συμφέροντα προς σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν πόλεμος γίνεται. Έχουμε μία παύση εχθροπραξιών και έχουμε μία θηρίδα που θα μας επιτρέψει να μπορούμε να παραδίδουμε ανθρωπιστική βοήθεια, να προσφέρουμε κάποια ελπίδα στους Σύριους και ένας από εσάς είπε πως, θα πρέπει να κάνουμε την απογοήτευση ελπίδα την απελπισία ελπίδα, έχετε δίκιο. Και να γεφυρώσουμε τα χάσματα μεταξύ των βασικών παικτών, να δούμε ποιο είναι ο κοινό τόπο και αυτή είναι η Ευρώπη και το πνεύμα της. Καμιά φορά αυτό δυσκολευόμαστε να το κάνουμε και στο εσωτερικό μας και καμιά φορά στο εξωτερικό τα καταφέρνουμε κάπως. Εν πάση περιπτώσει. Θα πρέπει να χτίσουμε το μονοπάτι για την ειρήνη, για την πολιτική αλλαγή στην ε, Συρία και να τους δώσουμε ένα μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο θα είναι δικό τους. Και δεν μιλώ μόνο για τους Σύριους που ζουν ακόμα στη χώρα, αλλά και για αυτούς που την έχουν εγκαταλείψει. Γιατί και αυτοί θα πρέπει να έχουν λόγο και για το παρόν και για το μέλλον της χώρας τους. Άρα λοιπόν πρέπει να πιέσουμε όλους τους παίκτες να μείνουν στα πλαίσια του οδικού χάρτη. Και για πρώτη φορά έχουμε και μία ένα ψήφισμα του ΟΕΕ που ε, εγκρίθηκε ομόφωνα. Και αυτό είναι το πολύτιμο αποτέλεσμα της δύσκολης δουλειάς που κάναμε. Άκουσα και κάποια λόγια για την έλλειψη ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε μου ξεκάθαρα, ε, επιτρέψτε μου να σας πω ξεκάθαρα πως εγώ ε, συμμετέχω σε πέντε διαφορετικούς σχηματισμούς του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου. Είμαι στο συλλογικό όργανο των Επιτρόπων. Είμαι εδώ, στο Κοινοβούλιο. Εδώ βεβαίως έχετε διαφορετικές απόψεις ως πολιτικές ομάδες, αλλά για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο είναι ενωμένη, στις σκέψεις, στις, ε, στα λόγια αλλά και στις πράξεις. Κάθε εβδομάδα, κάθε τρεις-τέσσερις μέρες συντονίζουμε ε, τις πράξεις μας, τα μηνύματά μας, τη δουλειά μας κάθε μέρα στις διάφορες ομάδες ε, δράσης. Μην περιγράφετε εσείς ως μη ενωμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν θέματα στα οποία δεν είμαστε ενωμένοι, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα για τα οποία πολιτικά όλοι βρισκόμαστε σε ίδιο μήκος Ας το πούμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς για μας, πολύ δύσκολο θα το παραδεχτούν κάποιοι άλλοι. Στη Συρία σήμερα η δράση μας είναι ενωμένη. Τώρα, πιο συγκεκριμένα. Λίβανος η Ορδανία. Συμφωνώ 100% και ίσως παραπάνω πως υπάρχει ανάγκη να υπογραμμίσουμε όχι μόνο την οικονομική στήριξη που μπορούμε να προσφέρουμε, αλλά και τα όσα μπορούμε να πετύχουμε έτσι ώστε να είναι πιο ανθεκτικές οι κοινωνίες εκεί, να αντέξει το σύστημα και να συνεργαστούν σε αυτά τα πλαίσια. Εγώ θα πάω στο Λίβανο και στην Ορδανία σε δύο περίπου εβδομάδες, σε δέκα μέρες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή, είναι στη Διεθνή Ομάδα Στήριξη μαζί μα, συνεργαζόμαστε και με την Ιορδανία και με το Λίβανο εξαιρετικά, γιατί έχουμε του ίδιου στόχου. Δηλαδή, να βρούμε μία λύση για τον πόλεμο, για τη χώρα, έτσι ώστε να ξεπεράσει ε, αυτή τη φάση και να ειρηνεύσει. Λογοδοσία. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε προσπάθειες με τις μη κυβερνητικέ οργανώσει που δρούν επί τόπου. και είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε αργότερα με περισσότερε λεπτομέρειε, είτε στην Ολομέλεια είτε σε μια από τι επιτροπέ. Με χαρά θα το κάνω. Και να κλείσω με ένα στοιχείο. Πολλοί από εσά, ή μάλλον κάποιοι από εσά, μίλησαν για το ρόλο των γυναικών. Για τη συγκεκριμένη αυτή η μέρα. Και άλλες μέρες θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, αλλά η 8η Μαρτίου κατά κάποιο τρόπο συνδέεται και είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν λέμε πως ε, το μέλλον της Συρίας θα πρέπει να ανήκει σε όλους τους Σύριους, σε όλους τους πολίτες εντός και εκτός χώρας, βεβαίως και συμπεριλαμβάνουμε τις γυναίκες. Και όταν μιλάμε, και όχι μόνο εμείς, οικοδομούμε τη δυνατότητα η Συρία να γίνει ένα κοσμικό κράτος, αυτό έχει να κάνει και με τις προσδοκίες των γυναικών στη Συρία για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη χώρα τους. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, στηρίζουμε την καθημερινή τους δουλειά και εντός και εκτός Συρίας με τους Σύριους και ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι στηρίζει μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ε, ασχολούνται με τη χειραφέτηση των γυναικών. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο με βρίσκει, με, με ιδιαίτερα και λυπάμαι που θα τελειώσω έτσι. Ξέρετε πως το τραπέζι... Ε, στο τραπέζι της ομάδας δράσης είμαι η μόνη που κάθομαι και είμαι γυναίκα. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στη διπλωματία σε πολλά μέρη στον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κλείσω όμως και λίγο πιο αισιόδοξα, να σας πω πως ναι, όταν οι γυναίκε είναι και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά και στις ομάδες διαπραγματεύσεων, όπως κάναμε για τη συμφωνία με το Ιράν, καμιά φορά έχουμε καλύτερες πιθανότητες να χτίσουμε κάτι. Ίσως είμαστε πιο ρεαλίστριες. Ίσως είμαστε πιο πεισματάρες αλλά τελικά ε, καμιά φορά είμαστε αποτελεσματικέ. Ευχαριστούμε Αντιπρόεδρε Μογγερίνη για την ε, δήλωσή σας που αφορούσε την κατάσταση στη Σύρια και ευχαριστώ και όλους τους